Καλησπέρα κυρίες ε, και κύριοι. Αρχίζουμε. Θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι πολύ ιδιαίτερο για σήμερα το απόγευμα. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 191 θα εκλέξουμε πρόεδρο σήμερα το απόγευμα. Έχω σημειώσει εδώ πέρα τα ονόματα βάσει του άρθρου 187 έτσι όπως τα πρότειναν οι πολιτικές ομάδες. Ε, απαιτείται απαρτία και αυτή είναι η στιγμή τώρα λοιπόν για να έχουμε τους υποψηφίους. Οπότε οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων παρακαλώ να πούν τα ονόματα των υποψηφίων. Κύριε Φιγερέδο, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είχα ανακοινώσει και στους συντονιστές της συνεδρίασή μας, η ομάδα μου προτείνει το βουλευτή μας, το Μικαέλ Γκούσταψον, ως υποψήφιο πρόεδρο για την Επιτροπή μας και αντικαθιστώντας την συνάδελφο Εύα Μπρίτ Βέντσον. Όπως ξέρουμε, έπρεπε λόγω ασθενείας να διακόψει τη θητεία της, την άσκηση της θητείας της και ο Μικαέλ Γκούσταυσον είναι ο αντικαταστάτης της, αναπληρωτής από το ίδιο κόμμα ο οποίος έχει μεγάλη πείρα στη χώρα του. Μεγάλη πολιτική πείρα και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερως με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, την ισότητα των φίλων και όπως είναι γνωστό ότι συμβαίνει με το κόμμα της αριστεράς στην Σουηδία. Είναι γνωστό λοιπόν και για το κοινοβουλευτικό του έργο και για το έργο του, την προσφορά του σε επίπεδο εθνικό. Έτσι λοιπόν προτείνουμε στην Επιτροπή αυτή την υποψηφιότητα, ελπίζοντας ότι όλοι μπορούν να στηρίξουν τον υποψηφιό μας, τον Μίκαελ. Thank you very much for your... Ευχαριστούμε. Και άλλες πολιτικές ομάδες έχουν να προτείνουν υποψηφίους. Όχι, δεν υπάρχουν άλλοι από ό,τι βλέπω, οπότε ο κύριος ε, Γκόσταυσον έτσι ορίζεται στη θέση του Πρόεδρου. There is also one more announcement. Άλλη μια ανακοίνωση πρέπει να σας κάνω. Διαβοήσε εκλέξαμε τον νέο μας Πρόεδρο. έχει, δηλώσει, έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και του παραδίδω την Προεδρία. Eh, Καλησπέρα σε όλους και σας ε, ευχαριστώ που με κλέξατε στη θέση αυτή. Ευχαριστώ για τη διεξαγωγή της ε, Προεδρίας, την Αντιπρόεδρο και προσβλέπω σε καλή συνεργασία μαζί σας. Ελπίζω επίσης ότι θα έχουμε και καρποφόρες συζητήσεις μαζί και ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αποφάσεις. Τώρα, κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, έχω δουλέψει για την ισότητα μεταξύ των ε, δύο φύλων σε πολλούς χώρους, στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα πιο πρόσφατα, και σε τοπικό επίπεδο, στις τοπικές αρχές δηλαδή στη Σουηδία, αλλά και στην καθημερινή ζωή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Πάντα ήμουν υπέρ της ισότητας μεταξύ των δύο φίλων. Και όταν τα παιδιά ήταν μικρά, για παράδειγμα, εγώ βοηθούσα τη γυναίκα μου. Είχαμε αποφασίσει να μοιράσουμε τις δουλειές, να πάρουμε και οι δύο γονική άδεια, εναλλάξει, για να μπορέσουμε και οι δύο να βοηθήσουμε με τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που αναλαμβάνω το καθήκον αυτό στην Προεδρία της Επιτροπής. Χαίρομαι πάρα, ε, λυπούμε μάλλον πάρα πολύ που η κυρία Πρίτ Σβένσον δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη θητεία της και το λέω αυτό γιατί η Πρίτ Σβένσον είναι μια υπέροχη προσωπικότητα. Και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό δούλεψε για την Επιτροπή αυτή η ίδια βοήθησε πολύ, πολλές γυναίκες ολόκληρη την Ευρώπη. Θα συνεχίσω κι εγώ στον ίδιο δρόμο. Φιλοδοξία μου είναι να συνεχίσω το έργο της, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα εδώ στην Ευρώπη. Θα συνεχίσω τη δουλειά της Εύα Μπριτ Σφένσον. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει η βία σε βάρος των γυναικών, υπάρχει το θέμα ε, της άνησης αμοιβή όπου οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο, υπάρχουν διακρίσεις επίσης βάρος των γυναικών στους χώρους εργασίας, όλα αυτά τα θέματα, όπως ακόμα και το θέμα των κλιματικών αλλαγών, όλα αυτά και πώς θα συμπεριλάβουμε και τη διάσταση του φύλου στο περιβάλλον, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλω να δουλέψω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω τώρα, απλώ θέλω να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι και το γεγονός ότι είμαι άντρας και μάλιστα είμαι ο πρώτος άντρας που αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής αυτής. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για μένα προσωπικά αυτό δεν είναι τίποτα το περίεργο γιατί τα θέματα της ισότητας μεταξύ των δύο φίλων είναι θέματα που δεν είναι θέματα των γυναικών μόνο. Τα θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φίλων είναι θέμα δημοκρατίας και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για μια καλή ζωή. Κανένας από τους δύο δεν πρέπει να γίνεται θύμα διακρίσεων εξαιτίας του φίλου του. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και εγώ και άλλοι άντρες να αναλάβουμε τις ευθύνες μας υπέρ της ισότητας μεταξύ των δύο φίλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Mr. Chair, on behalf of the group. Πρόεδρε, εκ μέρους της Επιτροπής σας καλωσορίζουμε εδώ και αν με επιτρέπετε δεν είχα την ευκαιρία προηγουμένως να τοποθετηθώ για να δώσω προτεραιότητα στην ε, διαδικασία. Όμως δύο λόγια για να πω πόσο πολύτιμη ήταν η Εύα Μπρίτ Σπένσον με την παρουσία της σε αυτή την επιτροπή. Τώρα αναλάβατε τη θέση της σε αυτήν την επιτροπή. Έχει γίνει τόση δουλειά από την Εύα Μπρίτ Σπένσον που είναι πολύ καλή ευκαιρία να αναλαμβάνει κανείς την Προεδρία αυτής της Επιτροπής. Ο κύριος Γκούσταυσον είπε όταν το επεσήμαναν πόσο το σχέ έχει δουλέψει η κυρία Σβένσον. Ξέρετε, η κυρία Σβένσον η ίδια την τελευταία φορά τη συνάντησα μου ότι είναι πλεονέκτημα που είμαι άντρα. Μπορώ να, το, να τοποθετηθώ καλύτερα στα θέματα των γυναικών ω άντρα και ω ουδέτερο μέρο. Αυτό τα λέει όλα νομίζω για τη θέση που έχει η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών στο Κοινοβούλιο. Η Προεδρία του κυρίου Γκούσταυσον μπορεί να κάνει τη φωνή μα να ακουστεί ίσω καλύτερα σε αυτού του σκληρού αγώνε που πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε τόσα θέματα. Είναι λοιπόν μεγάλη μα χαρά να σα στηρίξουμε κι εμεί τη δική σα την προσπάθεια. Καλώ ήρθατε. Okay, now we're moving on to... uh, on the uh, uh, free chairs announcement. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θα περάσω στα Från ordförande och det har οι ανακοινώσει του Προέδρου και το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αύριο το πρωί έχουμε δύο συναντήσεις με μια άλλη επιτροπή, 9.30 κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα προβλήματα των γυναικών στην Κεντρική και Νότια Αμερική και συνεχεία στις 11 έχουμε τη δεύτερη συνεδρίαση Με Και θα συζητήσουμε προβλήματα αυτής της Επιτροπής. Και προχωρώ στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Ε, στα διάφορα υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Κάτι άλλο, καμία παρατήρηση. Λοιπόν, η δεύτερη κοινή συνεδρίαση ήταν με την Επιτροπή Λίμπερ, την Επιτροπή Λίμπερ, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, αύριο στις 12. Λοιπόν, σας ανέφερα τις δύο κοινέ συνεδριάσεις, 9.30 με τη, για τις γυναικοκτονίες στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και 12 κοινή συνεδρίαση Λίμπερ ΦΕΜ. Στις 11 ε, Οκτωβρίου το απόγευμα θα έχουμε μια δημόσια ακρόαση με θέμα γυναίκες και αλλαγή του κλίματος. 3 με 6,5, ε, επισημεί κάποιος να πάρει το λόγο η κυρία Τόμσον. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να σας δεχτούμε εδώ πλέον ως ε, εκλεγέντα πρόεδρο μετά τις εξελίξεις ε, που είχε η Εύα Πρίτ, ε, αυτά που συνέβησαν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλήσατε για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μην ξεχνάτε όμως ότι εδώ μιλάμε και για τα δικαιώματα των γυναικών. Αποτελεί και συστατικό του τίτλου μας και ιδίω για τη διάσταση του φίλου Μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και Γι' αυτό προσβλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να εργαστούμε στα θέματα αυτά. Επίσης, γυναίκες με ειδικέ ανάγκες. Ε, δεν είναι μόνο το θέμα των ε, αρνητικών διακρίσεων. Ε, στη χώρα μου, παραδείγματο χάρη, οι άντρες με ειδικέ ανάγκες μπορούν να ζητήσουν την υπηρεσία ε, εκδιδομένων γυναικών από το Δήμο. Ε, άρα λοιπόν οι κατάσταση γυναίκες και τους άνδρες ε, είναι πάρα πολύ διαφορετικοί όσον αφορά τις διακρίσεις. Σας είπα ένα τέτοιο παράδειγμα του τι συμβαίνει με τους άνδρες και τι δικαίωμα μπορεί ενδεχομένως να έχουν από το Δήμο τους. παρακαλώ λοιπόν και τη διάσταση του φίλου να τη συμπεριλάβετε. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα η Δανία απέκτησε μια νέα κυβέρνηση. Μετά από 16 μέρες διαπραγματεύσεων έχει μια νέα κυβέρνηση με 23 υπουργούς, 14 γυναίκες, 14 είναι γυναίκες, είναι συνασπισμός τριών κομμάτων και ένα από από τα κόμματα αποφάσισε να ονομάσει μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες. Έχουμε γυναίκα πρωθυπουργό και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Έλε Τόνι Σμιτ ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1999 μέχρι το 2004. Και αυτή η κυβέρνηση θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1η 2012. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο σας έργο. Προέρχεται από μια χώρα όπου η ισότητα είναι εδρεωμένη και στην πολιτική πρακτική και στην κοινωνική ζωή. Ε, υπάρχουν πράγματα όμως πολύ σημαντικά που θα ανακαλύψετε εδώ, τα οποία θα έχουν αξία ακόμη και για τη χώρα σας, τη Σουηδία. Ε, το Κοινοβούλιο της Σουηδίας ε, μαζί με συναδέλφους, ε, είδαμε πόσο είχαν εντυπωσιαστεί από τη δουλειά, τη συστηματική δουλειά που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ισότητα των Φύλων και την πολυδιάστατη δουλειά. Με αφορμή αυτό που είπε η κυρία Τόμψεν το επαναλαμβάνω, διότι ένα σημαντικός ρόλος σας είναι να προωθήσετε τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Ε, δηλαδή, τη διάσταση του φύλου και αυτά που αποφασίζουμε εμείς εδώ, πώς εντάσσονται σε άλλες επιτροπές εμείς κάνουμε, ε, εκδίδουμε εκτός από αυτοτελείς εισηγήσει και γνωμοδοτήσεις για θέματα που επεξεργάζονται άλλες επιτροπές. Ένας ρόλος σας λοιπόν θα είναι πώς θα παρακολουθήσετε και θα, και θα απαιτήσετε ε, την ε, ένταξή τους στις πολιτικές της Ένωσης και γι' αυτό υπάρχει και ένα δίκτυο αρμοδίων βουλευτών για την ισότητα σε κάθε επιτροπή της, ε, ε, σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή και αν θέλετε από τη σχετική μου πείρα είμαι 12 χρόνια μέλος αυτής της επιτροπής παράλληλα με άλλες μου δραστηριότητες και την ε, επιδίωξη της πολιτικής ισότητας ως και σε ένα, πλαίσιο, σε ένα μέρος της αντιπροεδρίας μου είχα και αυτή την αρμοδιότητα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ένα, κάτι που ζητούμε από εσά ιδιαίτερα είναι πώς θα ε, τονώσετε και πώς θα αξιοποιήσετε αυτό το δίκτυο αρμόδιων και υπεύθυνων για την ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, πολιτική, οικονομική πολιτική, μεταφορές, περιβάλλον, υγεία κτλ. Και επιτρέψτε μου και μένα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση ε, όπου η νέα κυβέρνηση στη Δανία έχει γυναίκα με την πρωθυπουργό της σημερινή πρωθυπουργό της Δανίας. Είμαστε τέσσερα χρόνια μαζί συνάδελφοι στην Επιτροπή ε, κοινωνικών Υποθέσεων ε, και πιστεύω το ότι έχουμε μια νέα, ε, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στη Δανία και τον πρώτο πρόεδρο άνδρα στην Επιτροπή τη δική μας δείχνει σήμερα πώς τα δύο φύλλα συνεργάζονται και αναδεικνύουν τη συμπληρωματικότητα και τον αγώνα για ίση εκπροσώπηση. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κούρμαϊ. Ευχαριστώ. Να θυμίσω σε, όλες, σε όλους τους συναδέλφους ότι έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θαυμάσια εμπειρία για το θέμα της διάστασης των φίλων στη συνεργασία με άνδρες. Είμαι πολύ ευτυχής που δρόμα σήμερα και θα είμαι πολύ ευτυχής να συνεργαστώ μαζί σας τους ερχόμενους μήνες. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Εύα έκανε μια θαυμάσια δουλειά διότι ήταν και είχε μια θαυμάσια ηγετική προσωπικότητα ε, βοηθούμενη βεβαίως και από τη Σαμπίν και όλοι οι συνάδελφοι εδώ που κάθονται γύρω-γύρω έχουν μια εξαιρετική εμπειρία από τη συνεργασία μαζί της. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή κατανομή εργασίας και συνεργασία μαζί με τη γραμματεία ε, και, και με τους άντρες και με τις γυναίκες στη γραμματεία. Όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, αυτό παίζει πάντοτε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή μας και πολλές φορές ε, συζητούμε με τους συντονιστές μας θέματα ισότητας ε, και με τους συντονιστές των άλλων επιτροπών. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ε, και ως στην Αντιπροεδρία δηλαδή είχαμε την Άννα Ζαμπόσκα η οποία ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στο παρελθόν και την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσουμε τα θέματα της διάστασης του φύλου. Και έχουμε προχωρήσει σημαντικά, έχουμε κάνει μερικά σημαντικά βήματα και είναι επίσης σημαντικό να μην χάσουμε αυτή την προοπτική από τα μάτια μας και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε τι γίνεται παράλληλα και με τις άλλες επιτροπές. Θα έλεγα να έχουμε πάντοτε τις κεραίες μας ευαίσθητες για το θέμα της διάστασης του φυλού. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Θα ε, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την βραχνή φωνή μου και να σας συγχαρώ μαζί με όλους τους άλλους προλαλήσαντες. Η εκλογή σας δείχνει ότι ε, έχουμε τώρα έναν άντρα πρόεδρο της Επιτροπής, όχι μόνο, αυτό δεν μας ενδιαφέρει μόνο από απόψεως φίλου, αλλά επειδή έχει και μία αξία ε, το γεγονός αυτό διότι δείχνει ότι θεωρούμε, ε, εφαρμόζουμε πρακτικά αυτό το οποίο πρεσβεύουμε, δηλαδή ισότητα μεταξύ των φύλων. Και πιστεύω ότι με τη φωνή τη δική σας θα έχουμε μια ευρύτερη διάσταση σε όλα αυτά τα θέματα ισότητας και φύλου. Ο κύριος Ρωμίλα. Και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω εκ μέρου τη ομάδα των Πρασίνων. Αντικαθιστώ την Μαρέγια Κορνέλισον, την συντονίστρια, η οποία πολύ σύντομα θα επιστρέψει, λείπει με άδεια μητρότητας ακριβώς. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμεί ω Επιτροπή είναι να συμπεριλάβουμε και όλε τι άλλε επιτροπέ στι συζητήσει μα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και η πιο δύσκολη δουλειά που θα έχετε να κάνετε. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε για να συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις μας και τους συναδέρφους από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Μεταξύ άλλων ευθυνών θα έχετε και τις εξής προκλήσεις. Να ηγηθείτε εδώ της Επιτροπής αυτής, πράγμα στο οποίο θα σας διευκολύσουμε, θα σας διευκολύνουμε πολύ. Το άλλο είναι να κάνετε τη φωνή της Επιτροπής μας να εισακουστεί, να ακουστεί πιο πέρα. Αυτό θα είναι πιο δύσκολο. Ελπίζω πάντως να καταφέρετε και τα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Βαρβάνου έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους των φιλελεύθερων. Δεν θα είναι εύκολη δουλειά να είσαστε πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, γιατί εμείς περιμένουμε από τον πρόεδρό μας να εκπροσωπήσετε στο υπόλοιπο σώμα του Κοινοβουλίου τα θέματα τα οποία εμάς μας ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα τα πιο συγκεκριμένα που συζητάμε τους τελευταίους μήνες και για τα οποία έχουμε διχαστεί πολύ με την ΛΥΜΠΕ όσον αφορά και το πακέτο των θυμάτων. Έτσι λοιπόν, μια από τις πρώτες δύσκολες δουλειές που θα έχετε να κάνετε εσείς είναι να συναντηθείτε με τον πρόεδρο της ΛΥΜΠΕ και να συζητήσετε για άλλη μια φορά τη δυνατότητα και δύο επιτροπές να συνεργαστούν βάσει του άρθρου 51 και ελπίζω ότι εσείς θα τα καταφέρετε καλύτερα να τον πείσετε για το ότι η δικιά μας Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ στη δουλειά αυτού του πακέτου και ότι η ΛΥΜΠΕ έχει περισσότερες ευκαιρίες να πετύχει εφόσον δεχτείτε δικιά μας συνεργασία για να ετοιμάσουμε μαζί μια πολύ καλή έκθεση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα προκληθείτε να κάνετε. Ελπίζω να μπορέσετε όντω να μας βοηθήσετε γιατί η υπόθεση θα πάει στη διάσκεψη των πρόεδρων. Και εγώ πιστεύω στην ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να λυθεί συναδερφικά το ζήτημα αντί να φτάσουμε για τελική απόφαση σε κάποιον ο οποίος θα είναι ο διαιτητής τελικά στην υπόθεση. Καλή επιτυχία λοιπόν και στη μελλοντική σας δουλειά. σε ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να σας συγχαρώ ή να σας εκφράσω τα συλληπιτήριά μου. Διότι έχω πάντοτε την εντύπωση ότι εάν κανείς θέλει να τιμωρήσει κάποιον, ο Θεός θέλει να τιμωρήσει κάποιον, τον κάνει πρόεδρο της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Εντάξει, θαυμάζω την τόλμη σας και το θάρρος σας, αλλά μπορείτε να στηριχθείτε σε μένα, που πιστεύω ότι είναι πολύ καλό επιτέλους να έχουμε άντρα πρόεδρο της Επιτροπής. Και αυτό είναι θέμα gender mainstreaming που δεν το έχουμε διασφαλίσει τόσο πολύ στην ίδια μας την Επιτροπή, ενώ το διεκδικούμε εκτός Επιτροπής. Μπορείτε λοιπόν να υπολογίζετε σε μένα για να μην γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το έργο που έχετε αναλάβει. Thanks for that. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ζητά κανείς άλλο στο λόγο. Η κυρία Φεγγερέιδου. Ε, Ευχαριστώ. Παρόλο που δική μας ήταν η πρόταση, εξ ονόματος της ομάδας μου, να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που εστήριξαν αυτή την ε, εκλογή και να ευχηθώ στον Πρόεδρό μας πολύ και καλή τύχη στο κοινό μας έργο. για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φίλων. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα με πολύ καλή προεδρία όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και με αυτό τα τελευταία λόγια θα ήθελα να ε, ολοκληρώσω την πρώτη μου συνεδρίαση ως πρόεδρος. Θα κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών.